Dear colleagues, please, we will start. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε αυτήν την ε, κοινή συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής Απασχόλησης και Δικαιωμάτων των Γυναικών για να συζητήσουμε την έκθεση που εκπονούμε από κοινού για τη δημιουργία συνθήκων στην αγορά εργασίας που να ευνοούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σήμερα, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Η κυρία Μάριαν Τίσεν, η Επίτροπος ε, θα είναι στην Επιτροπή Απασχόλησης από τις 3 μέχρι τις 16 και 45 για να συζητήσει για τον διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή και στα πλαίσια αυτά θα μιλήσει και για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Βεβαίως, ναι μεν είναι στην Επιτροπή Απασχόληση αυτή η συζήτηση, αλλά και τα μέλη της δικής μας Επιτροπής μπορούν να συμμετάσχουν. Νομίζω ότι και εμείς ε, έχουμε συνεδρίαση όμως το απόγευμα. Θα είναι δύσκολο λοιπόν. Ε, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά να είναι σε δύο διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα θέλουμε ακόμη λίγο χρόνο για να το επιτύχουμε. Η επόμενη κοινή συνεδρίαση που θα κάνουν οι δύο επιτροπές μας δεν θα γίνει τελικά ε, όπως είχε προβλεφθεί, αλλά θα είναι στις 16 Ιουνίου 9 με 10 μετά από αυτές τις ανακοινώσεις να περάσουμε στη συζήτηση για την έκθεση όπου θα πάρουν το λόγο πρώτα απ' όλα η εισηγήτρια της Επιτροπής Ασχόλησης και γυναικών οι δύο εισηγήτρες οι κυρίες Λισκεβίτσους και Ντανόκα και μετά θα κάνουμε μία ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Στόλα και τον κύριο Σερβόζ που μας τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστώ. Για να ξεκινήσουμε, χωρίς να χάσουμε περισσότερο χρόνο, να δώσω το λόγο στην κυρία Λίνκεβιτσιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσουμε αυτή την κοινή μας έκθεση. Έκθεση την οποία έχουν εκπονήσει δύο συγγήτρες από δύο διαφορετικές επιτροπές, την Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Και όπως είπατε το θέμα μας είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθήκων στην αγορά εργασίας για την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματική ζωής. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε δύο γενικούς διευθυντές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα μαζί μας. Το κοινό αυτό σχέδιο έκθεσης είναι η δική μας η συμβολή για το ζήτημα αυτό και αποτελεί απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον οδικό χάρτη που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει στην εξισορρόπηση επαγγελματική και προσωπική ζωή. Ιδίω για τι οικογένειε που έχουν παιδιά. Ξέρετε ότι το καλοκαίρι του 2015 ξεκίνησε η σχετική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε και στη γενικότερη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με του κοινωνικού εταίρου. Εκπονώντα και συντάσσοντα την έκθεση αυτή, θα είμαι και εμεί επαφή με κοινωνικού εταίρου, εκπροσώπου, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπροσώπους συνδεκαλιστικών οργανώσεων και όντως η ανταλλαγή αυτή απόψεων ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούσαμε πολλές διαφορετικές επικοδομητικές απόψεις, οι οποίες συνέβαλαν πάρα πολύ στη δημιουργία της έκθεσης αυτής. Μπορούμε όντως ακούγοντας τις ιδέες αυτές να αυξήσουμε την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, προσφέροντάς τους τις δυνατότητες να εξορροπήσουν επαγγελματική και προσωπική ζωή. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ευθύ αμέσω τα βασικά, βασικότερα στοιχεία της έκθεσης αυτής, εκπροσωπώντας κυρίως την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ισότητα των δύο φύλων και τον ισότιμο επιμερισμό των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε ως επιτοπλίστων είναι ότι το ζήτημα της εξορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι περισσότερο πρόβλημα των γυναικών, καθότι οι γυναίκες στα πλαίσια της οικογένειας φέρουν περισσότερες ευθύνες. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε νομοθετικό και μη νομοθετικό μέτρο προκειμένου να ενθαρρύνουμε τον ισότιμο αυτό επιμερισμό των οικογενειακών ευθυνών. Θα πρέπει να αλλάξουμε πραγματικά τις νοοτροπίες μας τη στάση που έχουμε στον τομέα αυτό και επομένως θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο και τους κοινωνικούς εταίρους και μέλη της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη διαφορετική κατάσταση που έχουμε από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και την βελτίωση, την καλύτερη ανταλλαγή των πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το άλλο ζήτημα το οποίο θίξαμε είναι το ζήτημα της άδεια μητρότητο. Και αναφερθήκαμε σε έναν οδικό χάρτη που θα πρέπει να ακολουθηθεί, που μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να έχει ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή όμω δυστυχώ δεν έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Τα μόνα απτά μέτρα τα οποία βλέπουμε είναι σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδο όμω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μία ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή και με τη βοήθεια λοιπόν τη άδεια μητρότητα. Ζητούμε λοιπόν την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπροσωπείται στη σημερινή μα συνεδρίαση, προκειμένου να παρουσιάσει πολύ σύντομα μία πρόταση οδηγίας για την άδεια μητρότητα και προκειμένου να πληρώνονται για όλη τη διάρκεια της άδειας αυτής οι γυναίκες. Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια άδεια για τα άτομα τα οποία αναλαμβάνουν τη φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούν πολύ πιο εύκολα οι γυναίκες, οι άνδρες να προσέχουν ηλικιωμένους, να φροντίζουν άτομα με αναπηρία ή ακόμα και τα παιδιά και παράλληλα να χαίρουν της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και να έχουν και μία αμοιβή κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής. Ζητάμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία πρόταση για την άδεια ε, πατρότητας, μία οδηγία για την άδεια πατρότητας όπου θα πρέπει να προβλέπεται μία περίοδος τουλάχιστον δύο εβδομάδων η οποία θα πρέπει προφανώ να αμείβεται. Και ζητάμε επίση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για τη γονική άδεια, και να επεκτείνει το ελάχιστο αμοιβόμενο, την ελάχιστη αμοιβόμενη περίοδο από 4 σε έξι μήνες. Αυτά είναι τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που κάνουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα τέσσερα νομοθετήματα τα οποία θέλουμε να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε πλέον στο ίμιση της νομοθετικής αυτής βουλευτικής θητείας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους την υλοποίηση των τεσσάρων αυτών σημαντικών νομοθετημάτων και να μπορέσουμε και εμείς να τα επεξεργαστούμε. Σε αυτό το σχέδιο λοιπόν έκθεσης δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της παροχής των κατάλληλων συνθήκων για την φροντίδα των παιδιών. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε ουσιαστικά τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους στόχους της Βαρκελόνης και να βελτιώσουν τις δυνατότητες που δίνονται στις οικογένειες να χρησιμοποιήσουν ποιοτική και ποιοτικέ μάλλον και προσιτέ υπηρεσίε φροντίδα και φύλαξη των παιδιών. Οι υπηρεσίε αυτέ, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι προσιτέ και ποιοτικέ. Και θα πρέπει να έχουμε ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη φροντίδα των παιδιών προσχολική ηλικίας, να έχουμε τους κατάλληλου βρεφονιπιακούς σταθμού κτλ. Οφείλουμε επίση όλοι από κοινού να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίε, φροντίδας και φύλαξη των παιδιών σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης, στην έκθεση αυτή τονίζουμε ότι θα πρέπει να αναφερθούμε επίση και στο ζήτημα της ε, φροντίδας ε, μελών της οικογένειας ή ε, εξαρτώμενων μελών. Αναφέρομαι για παράδειγμα σε ασθενείς, σε ηλικιωμένους. Πολύ συχνά είναι οι γυναίκες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα αυτή και βέβαια δεν αμείβονται ποτέ αναγκάζονται επίση να εγκαταλείψουν την εργασία του ή να απουσιάσουν για κάποια χρόνια από την εργασία του και προφανώ αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο έπειτα και στα συνταξιδοτικά του δικαιώματα. Ζητούμε λοιπόν μέσω τη έκθεση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο προκειμένου να έχουμε στα πλαίσια του εξαμήνου συγκεκριμένου στοχευμένου δείκτε όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προ εξαρτώμενα άτομα ή ηλικιωμένου και θα πρέπει οι δείκτες αυτοί να μοιάζουν με τους δείκτες της Βαρκελόνης. Και προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το σύστημα αυτό, ζητούμε παράλληλα από τη Eurostat και τη Eurofound να συλλέξουν τα κατάλληλα δεδομένα και να εκπονήσουν χρήσιμες μελέτες. Όσον αφορά τώρα τους δείκτες αυτούς καθεαυτούς, ιδίως όσον αφορά για τη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών και την φροντίδα των ηλικιωμένων, οι δείκτες αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί γιατί μόνο βάσει τέτοιων δικτών μπορούμε να λάβουμε καλές αποφάσεις. Πρέπει επίση να μιλήσουμε για την επιδεινόμενη δημογραφική κατάσταση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται μνήμα στο ζήτημα αυτό στην εκθεσή μας. Η κατάσταση αυτή ξέρω ότι χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά ποσοστά γεννητικότητα στα κράτη-μέλη και σε ορισμένα κράτη τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν συνεχή και δραστική μείωση. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν καταφέρουν οι γυναίκες να εξορροπήσουν επαγγελματική και προσωπική ζωή, τότε ουσιαστικά δεν έχουν και κανένα κίνητρο για να αποκτήσουν παιδιά. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα απαραίτητα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα προκειμένου να εξισορροπήσουμε και να συμφιλιώσουμε την επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Το σχέδιο λοιπόν αυτό έκθεση επίσης επικεντρώνεται επίσης και σε ένα άλλο ζήτημα. Στο ζήτημα του ελεύθερου ποιοτικού χρόνου, καθώς επίσης και της δυνατότητας αναψυχής για τις γυναίκες και ιδίω για τις μητέρες. Ξέρετε ότι ο χρόνος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί δίνει τη δυνατότητα για διάφορες δραστηριότητες να ψυχής αλλά και για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη ενός ανθρώπου. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει προγράμματα περαιτέρω κατάρτιση επιμόρφωσης ή μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο οι γυναίκες όσον αφορά την προσοχή της προσωπικής τους υγείας. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά οι γυναίκες δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με την υγεία τους και με την προσωπική τους ανάπτυξη ή να ασχοληθούν με διάφορα χόμπι, δραστηριότητες αναψυχής. Ξέρετε ότι πολύ συχνά οι γυναίκες μετά τη δουλειά πηγαίνουν στο σπίτι και εκεί συνεχίζουν ουσιαστικά να εργάζονται καθότι όπω σα είπα υπομίζονται περισσότερο τι οικογενειακέ ευθύνε σε σύγκριση με του άντρε. Έχουν ελάχιστο λοιπόν χρόνο για τον εαυτό του, και κατά αυτόν τον τρόπο επιδεινώνει το οποιαδήποτε προσπάθεια εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό τη ισορροπία επαγγελματική και προσωπική ζωή είναι πολύπλοκο, πολύ σχηδέ, έχει πολλέ διαφορετικέ διαστάσει και πτυχέ. Θα υποβάλουμε λοιπόν εμεί διάφορε τροπολογίε προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό κείμενο, σε ένα κείμενο το οποίο θα φέρει ένα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πρέπει να πάει βέβαια προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ολοκληρώνοντα, να σα πω ότι προκειμένου να εξορροπήσουμε επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή ζωή, δεν υπάρχει μία ενιαία μαγική λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλε τι περιπτώσει. Συνεπώ, κάθε άτομο πρέπει να ψάξει να βρει τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο μπορεί να εξισορροπήσει επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή ζωή είμαι πεπισμένη ότι εργαζόμενοι από κοινού θα καταφέρουμε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Προσβλέπω στις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ολοκληρώνω λοιπόν στο σημείο αυτό τουλάχιστον όσον αφορά την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και εξ ονόματος Επιτροπής Απασχόλησης θα μιλήσει η κυρία Σντάνοκα. Ευχαριστώ κυρία Λικεβίτσιος και όπως ήδη αναγγείλατε από πλευρά τη Επιτροπής ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών η κυρία Σντανόκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε η Βίλα Πλανκεβιτσιούτε, οργανώσαμε μια σειρά συναντήσεων με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι προτάσεις που έχετε μπροστά σα προέρχονται από διάφορες πηγές. Δυστυχώς, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου και διακόπη λόγω των τραγικών γεγονότων στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της ε, ζωής των πολιτών μας. Όσον αφορά την ε, εξισορρόπηση επαγγελματικής ε, και ιδιωτικής ζωής, Δεν εννοούμε μόνο τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μιλάμε για τα δικαιώματα του καθενός. Να έχει οικογενειακή και ιδιωτική ζωή και ε, να εκπληρεί τα οικογενειακά του καθήκοντα χωρίς αυτό να ε, μειώνει το επίπεδο διαβίωσης του, να μην αντιμετωπίζει ε, κοινωνικό αποκλεισμό ή να πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο να βρίσκεται με την οικογένειά του και να απειλείται από φτώχεια ή να ε, διατηρήσει ένα επίπεδο διαβίωσης ε, αγνοώντας ε, την οικογένειά του. Θα πρέπει ο συνδυασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου να διασφαλιστεί για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο δηλαδή για τους νέους πατέρες, τις νέες μητέρες και τους φροντιστές. Η αδιαμητρότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της έκθεσής μας. Η έκθεσή μας δεν περιορίζεται όμως το θέμα αυτό. Σε κάποια οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται κοντά στο παιδί τους ε, ήδη από την, ε, τις πρώτες μέρες ζωής ε, του μωρού επειδή δεν υπάρχει ε, πατρική άδεια. Και θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε κάθε οικογένεια να μπορεί να κάνει τις επιλογές της ώστε να μπορέσει να εξισορροπήσει καλύτερα τον επαγγελματικό και οικογενειακό βίο στη δική της περίπτωση. Η ελεύθερη επιλογή γενικά είναι πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο επισημαίνουμε στην έκθεσή μας. Μιλάμε για ευέλικτες θέσεις εργασίας, τηλεεργασία, ε, εργασία με μηνωμένο ε, ωράριο, καθώς και ευελιξία όσον αφορά την γονική άδεια. Σημαντικό είναι κάθε άτομο, κάθε οικογένεια να μπορεί να κάνει τις δικές του επιλογές για να βρει την βέλτιστη λύση για την εξισορρόπηση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Ε, οι φροντιστές ε, δυστυχώς ε, προστατεύονται πολύ λιγότερο από τους γονείς από νομοθετικής πλευράς. Πολύ συχνά είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να φροντίσει το παιδί. Αν υπάρχουν λοιπόν διευκολύνσεις για τη φροντίδα των παιδιών σε κάθε κράτος μέλος, αυτό θα είναι θετικό. Σε πολλά κράτη-μέλη η φροντίδα δεν παρέχεται από επαγγελματίε. Και σημαντικό είναι όχι μόνο η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών, αλλά να είναι ε, και σχετικά οικονομικές. Θα πρέπει να προωθήσουμε την σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών στην εξέβρεση λύσεων για την εξισορρόπηση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Εάν θέλουμε να πετύχουμε πραγματική ισότητα ανάμεσα ε, στα δύο φύλλα, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, χρησιμοποιούμε καλύτερε τις δεξιότητές μας και να βελτιώσουμε τις δημογραφικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ανάγκη να εξυγχρονιστεί η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να αντιμετωπίσουμε ελλείψεις ή ακόμα και έλλειψη νομοθεσίας σε κάποιους τομείς. Ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλιστεί για να έχουμε ε, ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού. Η τηλεεργασία, ευέλικτες θέσεις, ε, ώρες εργασίας ε, ή η μερική απασχόληση δεν θα πρέπει να επιβληθούν σε κανέναν, θα πρέπει όμως να υπάρχουν ως επιλογή από την νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, ώστε ο καθένας ε, να μπορεί να κάνει μια σωστή επιλογή όσον αφορά το ωράριο εργασίας. Θα πρέπει να επιλέξει κανείς δηλαδή τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στη δική του οικογένεια. Και αυτό ισχύει και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Ισχύει για τις νέες οικογένειες, ισχύει και για ηλικιωμένους ανθρώπους. Γενικά, το πιο σημαντικό που θα πρέπει να πετύχουν τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που αναφέρονται στην έκθεσή μας είναι ε, η καλή ποιότητα διαβίωσης και αυτό ε, δεν περιορίζεται στο εισόδημα. Παρότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο εισόδημα. Μιλάμε όμως ε, και για την σωματική και ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη και την ε, αυτονομία των ανθρώπων ε, σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία του σχεδίου έκθεσής μας που ήθελα να επισημάνω. Πολύ ευχαρίστω. Θα ακούσουμε παρατηρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τις παρατηρήσεις εκπροσώπων των διαφορών πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίας δανόκα για την παρουσίαση αυτή. Και τώρα, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δώσω το λόγο στον κύριο Σερβός, Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να αντιδράσω στην έκθεση αυτή και να σας μιλήσω για την εργασία που διεξάγεται αυτή τη στιγμή για την πρωτοβουλία, για την ισορροπία επαγγελματικού προσωπικού βίου. Χαιρετίζω την έκθεση αυτή, τη διάβασα και σημειώνω ότι σε πολλά θέματα συμμεριζόμεθα τις εκτιμήσεις ε, των εισηγητριών. Ιδιαίτερα σε τρία. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια που είναι και πρόκληση για να έχουμε ισότητα και στην απασχόληση και στην αμοιβή στα 28 κράτη-μέλη και ιδιαίτερα σε εκείνα όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες. Δεύτερον, είναι σημαντικός αυτός ο συνδυασμός επαγγελματικής προσωπικής ζωής ούτως ώστε να συμμετάσχουν περισσότερο οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Και εμείς το καταλαβαίνουμε. Και επίσης σημειώνω ότι και οι πατέρες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στις οικογενειακές ευθύνες. Γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και νομίζω ότι το έχει τονίσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο. Τέλος, η σημασία ποιοτική φροντίδας για τα παιδιά και της ε, μακροχρόνιας φροντίδας για τα άτομα που τη χρειάζονται. Και αυτό το αναγνωρίζουμε. Η έκθεση λοιπόν αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρξει μια νέα προώθηση του θέματος αυτού και αποφασίσαμε να αποσύρουμε την οδηγία για την ε, άδεια μητρότητας πέρυσι. Και αυτό το κάναμε γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε μια ευρύτερη προσέγγιση για αυτήν την ε, ισορροπία και το συνδυασμό και γι' αυτό εκπονούμε τώρα την πρότασή μας ε, δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες αλλά θα αναφερθώ σε μερικά κύρια σημεία η Επιτροπή θα πρέπει να πάρει ως ε, συλλογικό σώμα την απόφαση αλλά γενικά νομίζω ότι και εμείς ασχολούμεθα με τα θέματα που κι εσείς κυρίως τονίζετε στις εκθέσεις. Να αναφέρω μερικά στοιχεία. Είναι πάντα σημαντικό. Το 14. Η απασχόληση των γυναικών στην Ένωση ήταν 63,4%. Ενώ για τους άνδρες ήταν 75%. Είναι πάνω από 10 εκατοστιαίες μονάδες ε, το χάσμα. Και αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι το 2006, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση, τα αντίστοιχα στοιχεία ήταν για τις γυναίκες 62%, 62,2% συγκεκριμένα. Δηλαδή από το 6% μέχρι το 16% δεν άλλαξε τίποτα. Δεν βελτιώθηκε η κατάσταση γιατί παρόμοια είναι τα ποσοστά. Ανησυχητικό ιδιαίτερα. Κάτι άλλο. Η Ένωση είναι σαφώς κάτω όσον αφορά το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών ε, από άλλες αναπτυγμένες χώρες. Στην Ελβετία, είναι πάνω από 77% η απασχόληση των γυναικών. Πάνω από 77% στην Ιαπωνία, 67% στις Ηνωμένε Πολιτείες, σχεδόν 71%. Άρα ε, είμαστε ουραγοί. Άρα υπάρχει ανάγκη να αναλάβουμε δράση για να βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και για να υπάρξει αυτή η ισορροπία γιατί αυτή η ισορροπία είναι βασικό στοιχείο για να βελτιωθεί η εργασία των γυναικών. Το ποσοστό εργασίας. Τώρα, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και μετά ίσως να πω και δύο λόγια για το περιεχόμενο της πρότασης που εκπονούμε. Για τη διαδικασία. Αξέρετε ότι ξεκινήσαμε την ε, πρώτη φάση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τον περασμένο Νοέμβριο. Ε, γιατί το κάνουμε αυτό για την νομική βάση είναι το άρθρο 153 της συνθήκης, όπου αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρξει μία πρώτη και δεύτερη φάση διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων. Και κατόπιν οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να αποφασίσουν να κάνουν διαπραγμάτευση για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των. Το 2010 για παράδειγμα το έκαναν αυτό και υπήρξε συμφωνία για τη γονική άδεια. Άρα έχουν εμπλακεί όλα αυτά τα χρόνια πολύ ενεργά στην εξέταση αυτού του θέματος και ελπίζω να καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η διαβούλευση και ελπίζουμε να καταλήξει θετικά. Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης φάσης της διαβούλευσης. Συνολικά σημειώνω ότι υπήρξε συμφωνία και από τις δύο πλευρές, εργαζόμενοι και εργοδότες, για την ανάγκη να υπάρξει δράση για να βελτιωθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και για την ανάγκη να βελτιωθεί η ισορροπία αυτή. Συμφωνούμε λοιπόν επί των στόχων. Ωστόσο, και εδώ προκύπτουν δυσχέρειες, δεν υπάρχει συμφωνία για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Οι εργοδότες, συγγνώμη, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, θα ήθελαν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και το είπαν ε, πολύ σαφώς ότι πρέπει να υπάρξουν νομοθετικέ πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα αυτά που αναφέραμε. Όμως από την πλευρά των εργοδοτών, η Business Europe και οι άλλε οργανώσεις δεν ενδιαφέρονται για νέε τέτοιε νομοθετικέ ενέργειε. Θεωρούν ότι η υπάρχουσα νομοθεσία είναι επαρκή και ότι είναι περισσότερο θέμα καλύτερη εφαρμογή τη υπάρχουσα νομοθεσία και ότι δεν χρειάζονται νέα νομοθετήματα. Βέβαια δεν θα αποφασιστεί τίποτα μέχρι να υπάρξει και η δεύτερη ε, φάση της διαβούλευσης. Σε αυτή τη δεύτερη φάση και οι δύο πλευρές, εργαζόμενοι εργοδότες, θα αποφασίσουν εάν θα διαπραγματευτούν μεταξύ των. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι αρνητική η απόλυξη της πρώτης φάσης. Αυτά που αναφέρουν οι εργοδότες στο σχετικό έγγραφο, να δούμε πώς θα αντιδράσουν στη δεύτερη φάση. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε το κείμενο που θα ξεκινήσει τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης. Ιδιαίτερα εκπονούμε ένα αναλυτικό κείμενο και είμαστε στην τελική φάση ε, εκπόνησης όπου τονίζουμε ποιες είναι οι αρχές της δεύτερης φάσης διαβούλευσης. Και μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση μας λοιπόν αυτή θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση. Και παράλληλα έχουμε ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση γιατί είναι σημαντικό να γίνει παράλληλα για να κερδίσουμε και χρόνο. Και θα σας εξηγήσει τι, να, τι είναι αυτή η δημόσια διαβούλευση που είναι ευρύτερη από τα θέματα που ανέφερα. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν σε φάση εκείνης της δεύτερης φάσης που είναι τμήμα του προγράμματος εργασίας μας για το 2016, άρα θέλουμε να ολοκληρωθεί στο μέτρο του δυνατού μέχρι τέλος του χρόνου. Τώρα δύο λόγια για το περιεχόμενο. Είπαμε ήδη ότι συμμεριζόμεθα την ανάλυση των εισηγητριών για τα κυριότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δύο λόγια για τα θέματα που εξετάζουμε. Δεν λέω ότι θα υπάρξουν νομοθετήματα από αυτόν. Απλώς αναφέρω τα θέματα που εξετάζουμε. Και θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι και μετά η Επιτροπή να αποφασίσουν εάν θα υπάρξουν νομοθετήματα επί κάποιων των θεμάτων που θα αναφέρω. Πρώτο θέμα. Άδεια μητρότητας. Σε τι επίπεδο και η διάρκεια. Προστασία κατά της απόλυσης μετά την άδεια μητρότητας. Πολύ σημαντικό θέμα. Και επίσης το θέμα των δυνατοτήτων και των διευκολύνσεων για το θυλασμό. <clears throat> και εξετάζουμε και το θέμα της άδεια πατρότητας. Όπως ξέρετε δεν υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία από αυτού μέχρι στιγμής και επανεξετάζουμε το θέμα της γονικής άδειας, επί των οποίων κοινωνική κοινωνικοί κατέληξε κατέληξαν συμφωνία το 2010. Αυτό καλύπτει όλα τα θέματα, αμοιβή, διάρκεια και επίσης ευελιξία. Για παράδειγμα, επιλογή ή όχι η γονική άδεια να γίνεται με μερική απασχόληση ή όχι. Επίσης εξετάζουμε τις μορφές απασχόλησης, να υπάρξει ε, ευελιξία για αυτούς που παρέχουν φροντίδα, για τις οικογένειες μέσω της χρήσης ε, τηλεεργασίας ε, ή ευέλικτων ωραρίων ή μερικής εργασίας για να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στους γονείς. Και κάτι που είναι σημαντικό για τις επιτροπές σας, εξετάζουμε το θέμα της ε, άδεια ε, χωρίς αμοιβή της ε, άνευ αποδοχών για να υπάρξει φροντίδα για κάποιους. Σας αναφέρω λοιπόν τα θέματα που μας απασχολούν, τα κύρια θέματα. Θα τα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει τις αποφάσεις της μετά τη διαμόρφωση άποψης των κοινωνικών εταίρων. Και να το συνδυάσω με την εργασία για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου τη διαβούλευση για τις αρχές του κοινωνικού πυλώνα. Μία από τις αρχές αφορά ακριβώς την ισορροπία αυτή, το συνδυασμό επαγγελματικής προσωπικής ζωής. Είναι σημαντική λοιπόν και διεξάγεται παραλίλου και αυτή η διαβούλευση, η διαβούλευση συγγνώμη, και να δώσω τώρα το λόγο στην Τίνα για να συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σερβός. Πριν τώρα να δώσω το λόγο στη συζήτηση με τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους ευρωβουλευτές και για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα παρουσίασης να δώσω το λόγο στην κυρία Στόλα που είναι Γενική Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση ε, Νομικών ε, Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τις δύο συγγήτριες, Μπλινκεβιτσούτε και Στανόκα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να βρίσκουμε εδώ πέρα σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία που αναλάβατε και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να έχουμε αυτή την κοινή συζήτηση σήμερα εδώ. Προφανώς θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να προωθήσουμε περισσότερο το ζήτημα της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ενδεχομένως να επαναλάβω κάποια από τα πράγματα που έχετε ήδη πει εδώ στην Επιτροπή σας, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και θετικό αυτό, γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι ε, σκεφτόμαστε και προσεγγίζουμε τον ίδιο τρόπο τα ίδια ζητήματα. Να αφαιρθώ καταρχάς στους γενικούς μας στόχους και στη συνέχεια θα αναφερθώ σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία ήδη έχετε αναφέρει εδώ στην Επιτροπή σας. Άδεια, δυνατότητα φροντίδας, ευελιξία, και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια διαβούλευση. Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμεριζόμαστε πολλά από τα ζητήματα τα οποία θίγεται στο σχέδιο έκθεσή σας και τα προσεγγίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα να τονίσω ένα συγκεκριμένο σημείο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τη νέα αυτή πρωτοβουλία και για την ισότητα των δύο φύλων. Αναφέρομαι στο ότι οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν αμοιβαία ισότιμη στάση ως εργαζόμενοι, αλλά και ο πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε αδικία και ανισορροπία υπάρχει όσον αφορά την έμιστη και αμοιβόμενη εργασία και να δούμε επίσης πώς μπορούμε να επιμερίσουμε καλύτερα τις οικογενειακές ευθύνες και τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων ανάμεσα σε άνδρε και γυναίκες. Το ζήτημα λοιπόν δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, είναι πολύ πιο ευρύ. Είμαι επίσης πεπισμένη ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το ζήτημα της μη αμοιβόμενη εργασίας, αλλά και με το ζήτημα της αμοιβόμενη εργασίας. Αν αφήσουμε το ένα από τα δύο ζητήματα, τότε η λύση που θα προτείνουμε δεν θα είναι ικανοποιητική. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στις γυναίκες κάθε φορά που συζητάμε τα ζητήματα αυτά, αλλά να δούμε και την περίπτωση των ανδρών. Δεν θα αναλύσω τώρα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας παρέθεσε ήδη ο κύριος Σερβός. Πάντως θα πρέπει να πω ότι θέλουμε και εμείς μια πιο ολιστική σφαιρική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το γενικότερο ζήτημα της εξορρόπησης επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Έχουμε ήδη ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, έχουμε ήδη συγκεκριμένα ευρωπαϊκά μέσα, έχουμε κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την πολιτική, αλλά όλα αυτά δεν αρκούν. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και θα πρέπει όλοι να συντοπίσουμε ποιο είναι το δυναμικό και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες στα πλαίσια της αγοράς εργασίας και πώς μπορούν να βρουν οι εργοδότες απαραίτητες δεξιότητες στα πλαίσια της αγοράς εργασίας, δεξιότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν ανάμεσα στο γυναικείο πληθυσμό εξετάσουμε λοιπόν ένα πακέτο μέτρων που θα περιλαμβάνει τόσο νομοθετικά όσο και μη νομοθετικά μέτρα. Η παροχή φροντίδας, οι, οι οικογενειακές ευθύνες είναι ένα γενικότερο ζήτημα το οποίο δεν θα πρέπει να βαρύνει μόνο τις γυναίκες προφανώς. Η πρόσβαση λοιπόν των γυναικών στην αγορά εργασία θα πρέπει να συνδέεται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στι οικογενικές υποχρεώσει. Και ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άντρε οι οποίοι θα ήθελαν να μπορούν να περνάνε περισσότερο χρόνο με τι οικογένειέ του. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα το ζήτημα των αδειών. Όσον αφορά την άδεια πατρότητας και την άδεια τη γονική, θέλουμε να έχουμε οδηγίες και για τα δύο αυτά ζητήματα, προκειμένου να δίνουμε περισσότερες επιλογές σε άντρες και γυναίκες, προκειμένου οι οικογένειες να μπορούν να πραγματικά να επιμερίζονται τις ευθύνες τους με τρόπο πολύ πιο εύκολο. Ο αριθμός των ανδρών που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε προτινόμενη γονική άδεια είναι πολύ χαμηλός. Έχουμε αυξητικέ τάσει σε κάποιες χώρες, αλλά γενικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όταν οι άνδρες, οι πατέρες χρησιμοποιούν τη γονική άδεια, αυτό το κάνουν για μια περίοδο πολύ πιο μικρή από ότι γυναίκες. Και επίσης, αυτό δεν μπορεί να οφείλεται μόνο σε καθαρά δική τους προσωπική επιλογή. Υπάρχουν σαφώς και διαρθρωτικοί λόγοι που επηρεάζουν την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε κάποια νέα μέσα τα οποία θα ενθαρρύνουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες να χρησιμοποιούν περισσότερο τη γονική άδεια. Πρέπει επίσης να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα την άδεια μητρότητας προκειμένου να υποφελούνται από αυτήν οι γυναίκες αλλά και να μπορούν να επιστρέφουν γρήγορα στην ε, αγορά εργασίας. Και ο κύριος ε, Σερβός Αναφέρθηκε επίση στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλέ φορέ οι γυναίκε στην επαγγελματική του ευδρομία όταν έχουν χρησιμοποιήσει μια άδεια μητρότητα. Τώρα, όσον αφορά τι υπηρεσίε παροχή φροντίδα, ξέρουμε ότι το ζήτημα τη εξορρόπηση επαγγελματική και προσωπική ζωή δεν ολοκληρώνεται μόνο με τη γέννηση του παιδιού ή με τα χρόνια εκείνα κατά την οποία το παιδί βρίσκεται σε νημπιακή ηλικία, τότε ξεκινάνε οι πραγματικέ ευθύνε και τότε πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει επιμερισμό των ευθυνών ανδρών και γυναικών, ιδίω όσον αφορά την φροντίδα των πολύ μικρών παιδιών. Θέλουμε λοιπόν εδώ πέρα να προωθήσουμε κάποια μη νομοθετικά μέτρα στα πλαίσια της γενικότερης δέσμης μέτρων και να καλύψουμε διάφορα ζητήματα, όπως το πόσο προσιτές και διαθέσιμες είναι οι υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης των παιδιών και πώς μπορούμε να καταρρύψουμε οποιαδήποτε αρνητικά κίνητρα μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών και τα οποία λειτουργούν πολλές φορές αρνητικά για τους άνδρες ή για τις γυναίκες. Σε 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολύ λιγότερες ε, θέσεις ε, σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ε, από ότι είναι η γενικότερη ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τις οικογένειες και να μην τις αφήνουμε μόνες τους και εκτεθειμένες στην επίλυση του προβλήματος αυτού. Στην έκθεσή μας στην εκθεσή σας, με συγχωρείτε, λέτε ότι θα πρέπει μέχρι το 2020 τα κράτη-μέλη να επιτύχουν τους στόχους της Βαρκελόνης. Και εμεί αυτό προωθούμε ω στόχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε επίση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κατάλληλο μέσο για να πετύχουμε την εξορρόπηση επαγγελματική και προσωπική ζωή. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τη φροντίδα των παιδιών, έχουμε χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σχετικού δείκτε και θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε και τα επόμενα χρόνια. Προτείνουμε συγκεκριμένα να συστήσουμε προς 10 κράτη-μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και γενικότερα να βελτιώσουν τους δείκτες ισότητας ανδρών και γυναικών. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της παροχής προσιτής φροντίδας των παιδιών. Το ζήτημα της ευελιξίας. Τώρα, οι εργαζόμενοι γονείς χρειάζονται ένα βαθμό ευελιξίας προκειμένου να καταφέρουν να οργανώσουν το εργασιακό και γενικότερα το πρόγραμμά τους κατά την περίοδο εκείνη που το παιδί είναι μικρό αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις ευελιξίας, αλλά σε εμβριακή ακόμα μορφή θα έλεγα, στα πλαίσια της οδηγίας για την γονική άδεια και προβλέπεται μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν υποφεληθεί της άδεια αυτής ή προβλέπεται για την περίοδο εκείνη που επιστρέφουν στη θέση απασχολήσή τους. Ορισμένοι τώρα εργοδότες προσφέρουν μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας και στους δύο γονείς, αλλά και πάλι στην ε, περίπτωση αυτή οι διευθετήσεις αυτές υπάρχουν μόνο για τους πλήρως απασχολουμένους. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μορφές εργασίας έχουν αλλάξει και λόγω της τεχνολογίας. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές οι γονείς και κυρίως οι γυναίκες αναγκάζουν να καταλήψουν την αγορά της εργασίας ή να απασχολούνται τελικά μόνο σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης που απαιτούν χαμηλή δίκευση. Πρέπει λοιπόν και αυτό το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι ε, οι γυναίκες είναι εγκλωβισμένες πραγματικά σε συνθήκες μερικής απασχόλησης και αυτό αργά ή γρήγορα τις οδηγεί σε πολύ υποδέστερη θέση όσον αφορά τις συντάξεις τους. Και πολύ συχνά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα 40% της τάξης 40% όσον αφορά τις συνταξιδοτικές αποδοχές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Επίσης έχουμε στατιστικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευελιξία χωρίς να αλλάξουν το εργασιακό του ωράριο ή χωρίς να επηρεάζει το συνολικό αριθμό ωρών που εργάζονται. Είναι οι γυναίκες αυτές οι οποίες αναγκάζονται να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους. Περίπου το 40% των γυναικών με παιδιά εργάζονται σε συνθήκε μερική απασχόληση, το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο για τους άνδρες. Πάντως, οποιοδήποτε πέρα από τους γονείς μπορεί τελικά και εξαιτία γύρω του πληθυσμού να πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή του να παράσχει φροντίδες προς εξαρτώμενα μέλη ή α, ηλικιωμένους α, γονείς για παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς στα πλαίσια της αγοράς εργασίας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα μπορέσουν τελικά οι άνθρωποι αυτοί να διατηρήσουν και να συνεχίσουν να παρέχουν τις δεξιότητές τους στα πλαίσια της αγοράς εργασίας και για αυτούς και για τους φροντιστές δηλαδή Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Αναφερθήκαμε επίση και στη δημόσια διαβούλευση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω κάποια πράγματα. Θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα τη διαβούλευση αυτή πριν το καλοκαίρι, αλλά θα μπορούσα ήδη από τώρα να σα δώσω κάποιε πληροφορίε. Στόχο μα ήταν να συγκεντρώσουμε διαφορετικέ απόψει για διάφορα μη νομοθετικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πολιτική καθοδήγηση, καλύτερη παρακολούθηση, καλύτερη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων και καλύτερο επιμερισμό των βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν. Λάβαμε συμβολή από 230 περίπου οργανισμούς και από 560 άτομα τα οποία συμμετείχαν στη διαβούλευση αυτή. Οι περισσότεροι οργανισμοί, το 98% των οργανισμών αυτό, συμφωνούν με τον τρόπο που περιγράφουμε τις διάφορες προκλήσεις και ένα 77% των απαντήσεων λένε ότι όντως πρέπει να αναλυφθεί περισσότερη ευρωπαϊκή δράση για την εξορρόπηση επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Όσοι απάντησαν θεώρησαν ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη διαθεσιμότητα καθώς επίσης και στο πόσο προσιτές μπορεί να είναι αυτές οι υπηρεσίες φροντίδας και, στο, και στο ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πιο ευέλικτες μορφές εργασίας. Ορισμένοι είπαν ότι χρειάζεται καλύτερη καθοδήγηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια ενίσχυση της παρακολούθησης της προόδου που σημειώνουν τα κράτη-μέλη. Το 70% των συμμετεχόντων το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα, πιθανέ λύσεις. Όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση μας είπαν ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στις υπηρεσίες φροντίδα των παιδιών και στις υπηρεσίες φροντίδα των ηλικιωμένων, ότι θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένοι πόροι για το ζήτημα αυτό και ότι θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα στους εργοδότες προκειμένου να απαιτείται και από αυτούς μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Ολοκληρώνοντα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μα. Για κάθε άτομο το οποίο βγαίνει σύνταξη έχουμε τέσσερα άτομα που εργάζονται. Το 2060 όμως τα άτομα αυτά θα έχουν γίνει δύο. Επομένως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσουμε την πολύ σημαντική, ε, το πολύ σημαντικό δυναμικό που έχουμε στα πλαίσια του εργασικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ενισχύσουμε ισότιμα δικαιώματα και για τους άνδρες και για τις γυναίκες στα πλαίσια της αγοράς εργασίας αλλά και όσον αφορά τον επιμερισμό των οικογενειακών ευθυνών. Προσβλέπω τώρα σε μια πολύ οικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με εσάς στα πλαίσια της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Στόλα και μετά από αυτές τις παρεμβάσεις που νομίζω ότι μας βοήθησαν να αποκτήσουμε μια ευρύτερη γνώση του θέματος αυτού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τις παρεμβάσεις των συναδέλφων, να αρχίσουμε με τους σκιώδεις και κατόπιν θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, εφόσον το επιθυμούν. Πρώτον, η κυρία Σιμιένσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το σχέδιο κειμένου που αποτελεί εξαιρετική βάση για την περαιτέρω συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε τους διάφορους τρόπους ε, συνδυασμού του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο, από το οποίο θα εξαρτηθεί το μέλλον πολλών οικογενειών της Ευρώπης. Η δημογραφική κρίση στην Ευρώπη είναι μία από τις ε, σημαντικότερες πτυχές που βλέπουμε. Έχει μειωθεί ο αριθμός γεννήσεων σε κάθε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πέσει κάτω από το επίπεδο που είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί ο πληθυσμός. Και επίσης αυξάνεται η ηλικία των ε, γυναικών που γεννούν το πρώτο παιδί τους. Ε, είναι γύρω στα 30 χρόνια τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ε, ότι υπάρχει αυτή η τάση, το πρώτο παιδί να γεννιέται σε μεταγενέστερο σημείο στη ζωή της γυναίκας. Χρήσιμο θα ήταν να υπάρχει επίδομα για κάθε παιδί. Θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες λύσεις όμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζοντας βέβαια και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην θεωρήσουμε την ε, μητρότητα ε, ή την ιδιότητα του γονέα ως ε, εμπόδιο στην σταδιοδρομία. Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα αγωνικής άδεια που να διασφαλίζει στη γυναίκα ότι μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη θέση της. Θα πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε σωστά το χρόνο εργασίας και να προωθήσουμε τις καλές πρακτικές. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε και για τους φροντιστές των ηλικιωμένων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να γίνουν πολλά, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε γύρανση του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε σοβαρά την πολιτική μας για τους ηλικιωμένου. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική αυτή έκθεση και προσβλέπω σε επικοδομητικό διάλογο στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Σότροβα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω εκ μέρους της συναδέλφου Καρπέλτς που είναι ε, σκιώδης ε, για το ΕΛΚ στο θέμα αυτό. Εκφράζει λοιπόν ε, την υποστήριξή της για την δημιουργία ευνοϊκών συνθήκων στην αγορά εργασίας για τον συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Θέλει επίσης η κυρία Καρπέλτς να συγχαρεί τους δύο εισηγητές, διότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και για την Επιτροπή Γυναικών και για την Επιτροπή Απασχόλησης. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου είναι ένα από τα θέματα που συζητούμε περισσότερο. Είναι παράγοντα κλειδί για την ενδυνάμωση των γυναικών και από την άλλη μεριά παρέχει την βάση για τον ποιοτικό χρόνο που περνούμε με τις οικογένειές μας. Γι' αυτό η κυρία Γκασπέλς πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό ώστε να προωθήσουμε άδειε ή υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών. Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε επικοδομητική προσέγγιση και όχι να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα που ουσιαστικά ε, να απειλεί την κατάσταση και θα πρέπει να σεβαστούμε την ε, αρχή της επικουρικότητας. θα πρέπει να έχουμε μία βάση που να μπορεί να υποστηρίξει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Καθπέλς είναι υπέρ της ισότητας ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ΕΛΚ όμως ε, δεν μπορεί να στηρίξει την παράγραφο για συμπερίληψη πυλώνα για τα δύο φύλλα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα επικεντρωθούμε στην εισαγωγή περισσότερων ε, παραγράφων για τα δικαιώματα των γυναικών ε, σε θέματα απασχόλησης. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή τελική έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σότροβα για την Άλντε, η κυρία Μίλνα. Α, δεν είναι εδώ. Οπότε, από την Επιτροπή Απασχόλησης, ο κύριος Χέτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η εισαγωγή αυτής της έννοιας ε, είναι περίπλοκη. Και ακριβώς αυτή πολυπλοκότητα ε, αντικατοπτρίζεται στο κείμενο των εισηγητριών, οι οποίε όμω κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώ και συμφωνώ με την προσέγγιση του. Στι κοινωνίε ε, τη Ένωση μα είναι πολύ δύσκολο για τι γυναίκε να συνδυάσουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή. Επίσης είναι δύσκολο να βρούμε χρόνο για να αναπτυχθούμε ως άτομα, ως προσωπικότητα και για να έχουμε και κάποιες περιόδους αναψυχής. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλα τα αναγκαία για να βελτιωθεί η κατάσταση. Να δημιουργήσουμε τουλάχιστον μια θετική ατμόσφαιρα για να επιτυγχάνουμε αυτόν τον συνδυασμό γιατί η αρμονική ανάπτυξη του κάθε ατόμου πρέπει να είναι βασικός στόχος της κοινωνικής και της πολιτικής μας στον χώρο της απασχόλησης και η δυνατότητα να φροντίσουμε για τα παιδιά μας είναι πολύ σημαντική και για τους δύο γονείς να μπορούν να συμμετάσχουν. Είναι πολύ σημαντικό. Στην τελευταία ολομέλεια εγκρίναμε ένα ψήφισμα για την ε, γονική άδεια και θα θυμάστε τι συζητήσεις κάναμε σε αυτή την ε, ολομέλεια και τονίζω πόσο σημαντικό είναι ακριβώς να μπορούν και οι πατέρες να αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτές. Να μπορούν και εκείνοι να συμμετέχουν στην ανατροφή των παιδιών τους από την πολύ μικρή του ηλικία γιατί έτσι δημιουργείται πολύ στενότερος δεσμός και είναι πολύ σημαντικό επίσης οι γονείς να μοιράζονται αυτές τις ευθύνες και όσοι άλλοι φροντίζουν άτομα που το χρειάζονται πρέπει επίσης ε, να έχουν αυτή τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι ε, επίσης πρέπει να έχουν το χρόνο για να αναπτυχθούν να αποκτήσουν και περισσότερα επαγγελματικά προσόντα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε γιατί μας δίνει πολλές ε, δυνατότητες ευελιξίας στην εργασία. Το σχέδιο έκθεσης αποτελεί τα σχέδια έκθεσης, είναι καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Θα υποβάλω διάφορες τροπολογίες και προσβλέπω σε περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρικε είναι εδώ παρακαλώ. Παρακαλώ η κυρία, όχι ο κύριος Γκέρι. Ευχαριστώ. Καταρχάς να συγχαρώ τις συγγήτρες για τις, εισηγήσεις, για τις του. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί πολύ περισσότερο με αυτά τα θέματα των οικογενειών. Είναι ώρα να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγική για τις οικογένειες. Έχω όμως ορισμένα προβλήματα με τα κείμενα. Για παράδειγμα, λένε ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα ο συνδυασμός της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Προσέξτε γιατί αυτό μπορεί να γίνει παγίδα. Ε, πώς συνδυάζεται αυτό με το δικαίωμα για την οικογένεια. Θέλετε να υπάρχει ένα πακέτο για την ισορροπία αυτή. Εγώ θα έλεγα να προωθήσουμε καλύτερα μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ε, οικογένεια. Λέτε ότι πρέπει να μπορεί να αναπτύσσεται συνεχώς το άτομο. Καλύτερα να αναφερθείτε σε επίδομα για την ανατροφή των παιδιών. Όλοι ξέρουμε ότι οι γυναίκες επειδή ως μητέρες αλαμβάνουν το μεγαλύτερο βάρος της ανατροφής των παιδιών έχουν περισσότερες ανάγκες. Να τους δώσετε επίδομα λοιπόν για την ανατροφή. Κοιτάξτε, δεν είναι διακοπές των να παιδιά. Είναι επάγγελμα και για ορισμένους πλήρους απασχόλησης. Αναφέρεστε στην άδεια μητρότητας και στη γονική άδεια. Πόσες φορές πρέπει να σας πω εδώ. Σταματήστε με αυτές τις ε, μεταφράσεις. Ε, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα να θεωρούμε ότι είναι άδεια, άδεια, δηλαδή σαν να είναι διακοπές η γονική άδεια. Όχι, είναι ε, απασχόληση. Πρέπει λοιπόν να μην χρησιμοποιούμε ε, λοιπόν σωστούς, ε, λάθος όρους. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την επικουρικότητα. Τη γνωρίζει την επικουρικότητα. Το βασικό είναι να έχουμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα να έχουμε οικογένεια και να είμαστε γονείς. Και πρέπει καλύτερα να βοηθούμε τους γονείς. Κάθε μητέρα, κάθε πατέρας που θέλει να πάρει μια άδεια άνευ αποδοχών για να φροντίσει τα παιδιά του, να ανθρέψει τα παιδιά του, μαθαίνει πολλά και αυτά που μαθαίνει μπορεί κατόπιν να τα αξιοποιήσει και στην επαγγελματική του ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Βάνα. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τις δύο συγγήτριες πρώτα για τα σχέδια εκθέσεων που είναι καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Ιδιαίτερα για να αναπτυχθεί περισσότερο η κοινωνική Ευρώπη και για την ισότητα ανδρών και γυναικών, ιδιαίτερα στην αγορά εργασία. Και για να γίνει αυτό, αυτή η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική προσωπική ζωή είναι θεμελιώδης. Γι' αυτό εμείς οι πράσινοι θα θέλαμε να αναπτυχθεί περισσότερο το θέμα της πολιτικής για τις γυναίκες αυτές τις εκθέσεις. Ήδη αναφέρθηκε. Διότι οι γυναίκες από πολλές, φορές, από πολλές απόψεις επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μόνο θέμα στατιστικών. Οι γυναίκες αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο για τις ε, οικιακές εργασίες και για την ανατροφή των παιδιών που δεν, ε, δεν πληρώνεται και πολύ περισσότερο εργάζονται με μερική απασχόληση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για την ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς. Όταν συζητήσαμε για την ε, οδηγία για την γονική άδεια, είδαμε ότι υπάρχει ανισότητα στη κατανομή των δυνατοτήτων δηλαδή για άδεια άνευ αποδοχών. Και σε αυτό συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή. Βεβαίως ε, η λέξη άδεια για αυτού του είδους, ε, την, ε, αυτού του είδους την απουσία από την εργασία δεν είναι σωστή, δεν είναι άδεια. Θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για χρόνο που αφιερώνεται στην ανατροφή. Πολύ λίγοι άντρες μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν την δυνατότητα χρόνου άνευ αποδοχών. Πιστεύω ότι γενικά οι άντρες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην ανατροφή των παιδιών και να έχουν περισσότερες δυνατότητες για την προστασία της πατρότητας, για παράδειγμα, και για, την, για το χρόνο άνευ αποδοχών για ανατροφή. Πιστεύω όμως ότι οι εκθέσεις αυτές πηγαίνουν ε, παραπέρα από το νοδικό χάρτη της Κομισιόν, οπότε είναι καλό. Και είναι σημαντικό για μας να υπάρξει και ένα νομοθετικό κείμενο σε επίπεδο που να είναι το αντίστοιχο ε, με το χρόνο μητρότητα 24 εβδομάδε, για παράδειγμα, και να υπάρχει υποχρεωτική άδεια πατρότητα 2 εβδομάδων. Υποχρεωτική. Όπω είπαμε και για τη γονική άδεια. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ισότητα. Επίσης θα θέλαμε να υπάρχουν και περισσότερες αναφορές σε κίνητρα, ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα για τι γυναίκε, ώστε να, να μπορέσουν να, να επιστρέψουν στην εργασία. και θα θέλαμε να γίνει μία αναφορά και στις οικογένειες LGBTT. να υπάρχουν ε, ε να υπάρχει ισότητα και για αυτές τις οικογένειες για λεσβίες ε, φιλομεταβατικά άτομα κτλ να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να λαμβάνουν τέτοιες υπηρεσίες του επίπεδου είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη και για την εισηγήτρια από την Επιτροπή Γυναικών θέλω να τονίσω ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχει ευρύτερα η κοινωνία των πολιτών και των ελληνικών εταίρων ζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ η Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες όσον αφορά την έκθεση τους αυτή για την εξισορρόπηση επαγγελματική προσωπικής ζωής. Όσον αφορά τον τίτλο, θεωρώ ότι είναι σημαντικός. Έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάμε για συνδυασμό, συμφιλίωση, αναφερόμαστε μόνο στους γονείς. Αλλά δεν είναι μόνο οι γονείς αυτοί οι οποίοι πρέπει να συνδυάσουν επαγγελματική και προσωπική ζωή. Υπάρχουν απλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν και αυτή μία προσωπική ζωή, οι οποίοι δεν θα πρέπει να βρίσκονται μόνο στο γραφείο, αλλά θα, μπορούν, θα πρέπει να μπορούν να ζουν κανονικά και την ιδιωτική του ζωή. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην επηρεαζόμαστε μόνο στους γονείς. Θα πρέπει να εστιάσουμε καλύτερα στην εξορρόπηση επαγγελματική και προσωπικής ζωής για όλους. Το είπε και η συνάδελφος πριν από λίγο, ο συνδυασμός αυτός, η εξισορρόπηση αυτή ουσιαστικά αφορά περισσότερο τις γυναίκες, γιατί αυτές ακολουθούν περισσότερο ένα πιο παραδοσιακό ρόλο ανάληψης των οικογενειακών υποχρεώσεων, ακόμα και αν δεν είναι μητέρες αλλά και από στατιστικής πλευράς βλέπουμε ότι οι γυναίκες συμμετέχουν λιγότερο σε προγράμματα κατάρτισης εκτός εργασίας γιατί έχουν λιγότερο χρόνο τελικά και αυτό οδηγεί τελικά σε διακριτική μεταχείριση όσον αφορά και την ίδια τη δουλειά αλλά και την αναψυχή και τον εύθερο χρόνο. Πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να πετύχουμε εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για όλους και όχι μόνο για τους γονείς. Πρώτο ζήτημα, το χρονοδιάγραμμα το οποίο μας προτείνατε εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημόσια διαβούλευση. Προβλέπετε δημόσια διαβούλευση από τις συνθήκες. Πολύ καλά. Ακούσαμε ότι η Business Europe δεν θέλει πάρα πολύ να επεξεργαστούμε κάποιο νομοθετικό μέσο. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας επιτρέψει να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο προκειμένου η ε, εργαζόμενοι, οι ομάδες εκπροσώπησης των εργαζομένων να μπορούν να καταλήξουν τελικά σε μία απόφαση προκειμένου τελικά να έχουμε και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το 2017. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ κρίμα στα πλαίσια της προτινόμενης αυτής νομοθεσίας να μην έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις βάσω συγκεκριμένων πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνο και μόνο επειδή ένας από τους κοινωνικούς εταίρους δεν θέλει αυτή τη στιγμή νομοθετικά μέτρα. Η Επίτροπος Γιούροβα μας είπε στην Ολομέλεια ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αυτή η ίδια θα αναλάβει προσωπικά να προωθήσει μια πρωτοβουλία. Πρέπει να αναλυφθεί δράση. Επίσης, ξέρετε ότι από το 1996 έχουμε την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Έκτοτε τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν όσον αφορά τις συνθήκες ε, φροντίδας των παιδιών αλλά και τις εργασιακές συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένη πράξη αναθεώρησης οδηγίας αυτής. Θα μείνετε λοιπόν στο χρόνο χρονοδιαγραμμά σα ή θα επιτρέψετε περισσότερο χρόνο για την εξέλιξη αυτής της δημόσιας διαβούλευσης. Μας είπατε επίσης ότι θέλετε μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Μας δυσαρέσει το γεγονός ότι εγκαταλείψατε την άδεια μητρότητα, την αρχική πρόταση που είχε υποβληθεί, αλλά αποδεχόμαστε τις τάσεις γιατί μα είπατε ότι θέλετε να έχετε μια πιο ευρεία προσέγγιση. Έχουμε όμως και την άδεια πατρότητα και τη γονική άδεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε και τις τρεις αυτές προτάσεις να τις επεξεργαστούμε προκειμένου να ωφελήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα επηρεαστούν από τις άδειε αυτές. Όσον αφορά τη γονική άδεια, είδαμε ότι όταν δεν προβλέπεται μια άδεια πατρότητας, είναι πολύ δύσκολο και για τον ίδιο τον πατέρα να αποφεληθεί τελικά από τη γονική άδεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία ή αν μη τι άλλο για ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άδεια πατρότητας προκειμένου να μπορούν να υποφεληθούν για την περίοδο αυτή και οι ίδιοι οι πατέρες. Όσον αφορά την γονική άδεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τη διάρκεια, την αμοιβή και την μη μεταβιβασιμότητα των δικαιωμάτων αυτών. Επίσης, οι δομές υποδοχής. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δημόσιες τέτοιες δομές, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται και απαραίτητη πόρη, απαραίτητη χρηματοδότηση. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε εμείς να μπορούμε να έχουμε αυτούς τους περίφημους δείκτες στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι για μας σημαντικό γιατί ουσιαστικά μας επιτρέπει να παρακολουθούμε λίγο τις τάσεις στα κράτη-μέλη. Είναι κρίμα να, περιοριζόμαστε, να περιοριζόμαστε, με συγχωρείτε, μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε και κοινωνικούς δείκτες ή δείκτες σαν αυτούς που σας προτείναμε. Έπειτα, όσον αφορά την εγγύηση για τη φροντίδα των παιδιών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Child guarantee, να μπορούμε να προβλέψουμε κάτι συγκεκριμένο για τα παιδιά. Ήμουν χθε μια συνεδρίαση για την καταπολέμηση της ένδυας στα παιδιά. 22 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συνθήκες φτώχειας και αυτό διότι οι γονείς τους βασικά είναι φτωχοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό της ένδυας, το φαινόμενο της φτώχειας, το οποίο βέβαια συνδέεται με άλλα ζητήματα όπως ο ελάχιστος μισθός, οι ποιοτικέ δομές υποδοχής Πρέπει λοιπόν και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μπορούμε να παρακολουθούμε συστηματικά τους δείκτες αυτούς προκειμένου να μπορούμε να προτείνουμε έπειτα μεταρρυθμίσεις σχετικές και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Petit. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τις εισηγήτριες. λαμβάνονται βήματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Δεν έχουμε πετύχει το στόχο ακόμα όμως. Και μας ενδιαφέρει όχι μόνο η ευημερία των ατόμων, αλλά μας ενδιαφέρει και το όφελος για την κοινωνία γενικά, διότι είναι γνωστό ότι οι ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι και πιο παραγωγικοί εργαζόμενοι. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι η αμοιβή είναι το μόνο κίνητρο για τους εργαζόμενους και να υπάρχουν ε, τρόποι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει στην αγορά εργασίας με τον τρόπο που είναι καλύτερος για την ε, δική του ζωή. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας και οι λύσεις που συμβάλλουν στη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου βοηθούν την ένταξή του στην αγορά εργασία, για παράδειγμα η μείωση του ωραρίου ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά του ή άλλα μέλη τη οικογένεια. Και επίση είναι κάτι που επηρεάζει την ε, απόφασή του ε, για το πόσα παιδιά θα κάνουν, κάτι που ε, συνδέεται και με τι δημογραφικέ τάσει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. τα θέματα για την ε, φροντίδα των ε, γονέων ε, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 4. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών να μην είναι υποχρεωμένες να εργάζονται για τρεις εβδομάδες χωρίς, χωρίς άδεια ή κάποια μέρα εξεκούρασης. Ε, είναι θέματα που συνδέονται με πολύ άγχος και ψυχοσωματικές διαταραχές, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να αφιερώσουν χρόνο και στις οικογένειές τους. Μάλιστα, τον χρόνο που περνούν με τις οικογένειές τους είναι πολύ κουρασμένοι και ε, αφηρημένοι και κάτι... Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κακό για την οικογενειακή ζωή, καθώς και για το χρόνο που αφιερώνει κανείς για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Η ξεκούραση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά η αντικατάσταση άλλης μέρας ξεκούρασης δεν είναι ικανοποιητική λύση, καθότι ε, δεν ε, έχουν ε, ελεύθερη την κάποια άλλη μέρα στην εβδομάδα. Σημαντικό είναι λοιπόν οι οικογένειε να μπορούν να συγκεντρώνονται τι Κυριακέ, ε, για παράδειγμα. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να αναφέρετε ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίζονται ε, καλές ε, ώρες εργασίας και η μία μέρα ανάπαυσης να είναι η Κυριακή. Thank you. Ευχαριστώ. πολύ. Η κυρία Κοσλός Καράτοβιτς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τις εισηγήτριες και όλους όσους συμμετείχαν στην σύνταξη της έκθεσης αυτής. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλό έγγραφο, παρότι δεν συμφωνώ κατά 100%. Αποτελεί πολύ καλό έγγραφο και επικεντρώνεται στα βασικά σημεία ενός θέματος που είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Οι γυναίκες ε, μέχρι τώρα ε, έφεραν διπλά βάρη. Ε, θέλουμε να διατηρήσουμε τα καλά στοιχεία από την απελευθέρωση των γυναικών και από τη χειραφέτηση των γυναικών ε, και να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις δυσκολίες. Ε, λέμε ότι υπάρχει ένα χάσμα στην απασχόληση 10 ποσοστιαίων μονάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Ε, αλλά σημαντικό είναι και το 40% συνταξιδοτικό χάσμα που έχουμε. Οι γυναίκες ε, στην αγορά εργασίας ε, συχνά εργάζονται με μειωμένο ωράριο και έτσι οδηγούμαστε στο συνταξιδοτικό χάσμα. Συμφωνώ με τις εισηγήτριες ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται μέσα στην οικογένεια. Ο επιμερισμός των καθηκόντων μέσα στο, στην οικογένεια είναι πολύ σημαντικός. Διότι δεν μπορεί κανείς να πολλαπλασιάσει το χρόνο που περνά με την οικογένειά του. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ταυτόχρονα τις δουλειές του σπιτιού την ώρα που δουλεύουμε. Θα πρέπει όμως να παράσχουμε τρόπους ώστε να είναι πιο εύκολη η λήψη τέτοιων αποφάσεων εντός της οικογένειας. Κάποιοι εργοδότες θεωρούν ότι επιχειρηματική κουλτούρα είναι πιο σημαντική από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις ε, την ε, οικογένεια. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εξωσορόπηση ανάμεσα στον επαγγελματικό και τον οικογενειακό βίο. Νομίζω όμως ότι το κλειδί ε, δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια με μεμονωμένων επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να υπάρχει και σχετική νομοθεσία είναι απαραίτητη μια σειρά νομοθετικών λύσεων. Για παράδειγμα, έχουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στο σπίτι τους. Χρειαζόμαστε λύσεις όχι αποκλειστικά θεσμικού χαρακτήρα. Πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παράδοση που θεωρεί ότι κάποια πράγματα λύνονται καλύτερα εντός της οικογένειας, εντός του σπιτιού. Για παράδειγμα, η φροντίδα των ηλικιωμένων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλές ρυθμίσεις ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε τις οικογένειες διατηρώντας στο βαθμό που είναι δυνατόν το παραδοσιακό μοντέλο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει να υπάρχει ενιαίο καθεστώς για όλους τους φροντιστές, διότι υπάρχουν οποίοι φροντίζουν τα παιδιά, αλλά συχνά και τους ε, ηλικιωμένους. Ε, και μάλιστα και παιδιά και ηλικιωμένους ταυτόχρονα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ενιαίο καθεστώς για αυτούς τους φροντιστές και να έχουμε ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν ευέλικτες λύσεις για την πρόσληψη φροντιστών. Διάφορα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διάφορα μέσα, χρειάζεται όμως να έχουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τον τομέα αυτών και στην εκθεσία αυτή και στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, μου αρέσει η ιδέα να συμπεριληφθούν τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ώστε να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση και καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη. Και φτάνουμε στο πολύ σημαντικό θέμα της επικουρικότητας. Συμφωνώ ότι η γονική άδεια και η φροντίδα είναι θέματα επικουρικότητας. Χρειαζόμαστε μια νομική γνωμοδότηση ώστε να μην υπονομευθούν οι προτάσεις μας λόγω επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Thank you for intervention. Ε, Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που ήσασταν εδώ. Είχαμε σχόλια, είχαμε και ερωτήσεις. Κύριε Σέρβος, παρακαλώ. Από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση. Να πω κάποια πράγματα απαντώντα στι ερωτήσει. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω για τι ερωτήσει αυτέ, για τι παρατηρήσει σα. Βλέπω ότι σε πολλά σημεία συμφωνούμε. Στα όσα λέγονται δηλαδή στο σχέδιο έκθεση, στα όσα σα είπα πριν από λίγο και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά υπάρχει μια κοινή προσέγγιση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι απόψει που πρασβεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω δύο τρία πράγματα. Πρώτον, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κερδίσουμε και οι δύο. Είμαστε σε μια κατάσταση win-win όπως λέμε. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για την ισότητα από τη μία πλευρά, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά από την άλλη, από οικονομική κολλά πλευρά, το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ουσιαστικά συμβάλλουμε στην οικονομική ευημερία των κρατών μελών, αν υπάρχουν περισσότερε γυναίκε που θα συμμετέχουν στην αγορά εργασία. Ξέρετε ότι σε μορφωτικό επίπεδο υπερτερούν πλέον οι γυναίκες έναν των ανδρών. Παρ' όλα αυτά συμμετέχουν λιγότερο στην αγορά εργασίας. Αυτή την αντίφαση θα πρέπει να την επιλύσουμε. Και αν δούμε τα αριθμητικά δεδομένα ανάμεσα στα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν χαμηλά ποσοστά γεννητικότητα είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία έχουν τελικά και έναν ενεργό πληθυσμό που όλο και συρρυκνώνεται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό καθαρά από οικονομικής πλευράς να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Και βέβαια κερδίζουν και οι δύο πλευρές γιατί λύνοντας το οικονομικό αυτό πρόβλημα ωφελούμε και το ζήτημα της εξορρόπησης επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Και συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να ενταχθεί το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ήδη φύσταται γιατί στις συστάσεις που κάνουμε το καλοκαίρι αλλά και κάτι διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με ζητήματα ισότητας των φύλων που πρέπει να επιληθούν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Μάλτα, για παράδειγμα, σε σχέση με τις συζητήσεις που είχαμε εκεί, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δωρεάν παροχή υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά παντού στη χώρα αυτή. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Είναι ένα από τα μέσα που θα πρέπει, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε, αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεύτερον, όπως υπόθηκε ήδη, Πρέπει να βελτιώσουμε την ισορροπία επαγγελματική και προσωπική ζωή με τρόπο πιο γενικό και σφαιρικό. Προφανώ επικεντρωνόμαστε στου γονεί, αλλά συμφωνώ μαζί σα ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στου γονεί. Τα μέτρα τα οποία επεξεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν να κάνουν γενικά με την οργάνωση εργασία, με την ευελιξία που μπορεί να έχει κανεί για να κάνει τηλεεργασία, για να εργαστεί σε καθεστώ μερική απασχόληση και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να βελτιώσει και το επίπεδο εκπαίδευσής του, θα έχει περισσότερο χρόνο να ακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης κτλ. Όσον αφορά επίσης το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα ευνοϊκά για τους πατέρες. Συμφωνώ μαζί σας. Η κατάσταση θα βελτιωθεί όταν οι ίδιοι οι πατέρες αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την οικογένειά τους. Θα βελτιωθεί και η δική τους η κατάσταση στα πλαίσια της αγορά εργασίας. Να μπορεί να προβλέπονται δηλαδή περισσότερες δυνατότητες για να αφήσουν τη δουλειά τους εν μέρη και να ασχοληθούν λίγο με την οικογένειά τους όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα. Η πρόταση για την εξορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ε, αυτή τη στιγμή προβλέπεται στο φετινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί μέχρι το τέλος του έτους ή το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2017 θα πρέπει να ολοκληρώσει την πρότασή της. Άρα εμεί, απαντώντα στο ερώτημά σα, θα ακολουθήσουμε το αυστηρό αυτό χρονοδιάγραμμα που προτείναμε. Θα πρέπει να τηρήσουμε όμως τη διαδικασία που προβλέπεται από τις συνθήκες, θα περάσουν, όπω σα είπα πολύ σύντομα, στη δεύτερη φάση διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα έχουν στη διάθεσή του έξι εβδομάδες για να καταλήξουν σε μια απόφαση, αν οι εργοδότε πούνε τελικά ότι δεν ενδιαφέρονται για τη διαβούλευση αυτή, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε τη, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ήδη ότι θα υπάρξει μία δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων και αυτό αποτελεί τμήμα τη αρχική ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα εργασία τη το 2016. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα. Και τώρα η Τίνα Άστολα, Γενική, Διεύθυνση, Γενική Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Just. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, αλλά ίσως ορισμένα. Τώρα για τις άδειε, όπως υπόθηκε, δεν πρέπει κανείς να ηθικολογεί επ' αυτού. Συμφωνώ ότι εάν οι πατέρες πάρουν άδεια πατρότητας, κατόπιν μοιράζονται καλύτερα τα βάρη τροφής. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε συνολικά αυτά, ως πακέτο, και όχι απλώς να επιλέξουμε κάποια από αυτά. Αναφερθήκατε και υπήρξε απάντηση μάλιστα και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, με την οποία συμφωνώ. Το βασικό είναι βεβαίως να συλλέγουμε τα σωστά στοιχεία μέσω των σωστών δικτών και σε διάφορα ε, δικαστικά θέματα. Είναι πολύ βασικό να έχουμε τους σωστούς δείκτες για να μην καταλήγουμε σε λάθος συμπεράσματα. Και το βασικό είναι να μην ασχοληθούμε μόνο με νομοθετικά αλλά και με μη νομοθετικά θέματα. Αναφέρθηκε είναι θέμα νοοτροπίας αντιμετώπισης. Βεβαίως είναι θέμα νοοτροπίας εντός των οικογενειών, εντός των κοινωνιών, αλλά για να αλλάξουν οι νοοτροπίες πρέπει να υπάρξει και αλλαγή της δομής και ευαισθητοποίηση. Άρα τα κίνητρα και τα αντικίνητρα θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Λινκεβισούτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλους τους ομιλητές για τις προτάσεις τους, για τα σχόλιά τους. Να ευχαριστήσω βέβαια και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους, όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τις προτάσεις που έκαναν. Το έγγραφο που έχετε μπροστά σας είναι απλώς ένα σχέδιο εγγράφου. Αναμένουμε τις δικές σας προτάσεις, τις δικές σας τροπολογίες, προκειμένου να έχουμε μία ισχυρή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε σε κάθε περίπτωση ότι θα συζητήσουμε πολύ καλά τη θέση μας αυτή και ότι θα είναι και εύκολος εφαρμόσιμη στη συνέχεια. Κάποια σύντομα συμπεράσματα μετά τη σημερινή συζήτηση. Από ό,τι φαίνεται, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις, σε κάποιους τρόπους, προκειμένου να πετύχουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον καθένα μας. Είναι σημαντικό για τις οικογένειες, είναι σημαντικό για όσους δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν παιδιά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ακριβώς αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να επιλύσουμε. Αναφερόμενοι σε αυτά που είπε ο κύριος Σαββός για την διαβούλευση. Από ό,τι καταλαβαίνω και οι ίδιοι κοινωνικοί εταίροι βλέπουν ότι φύστε το πρόβλημα αυτό, ή την εργοδότες ή την εργαζόμενη απλώς διαφωνούν ως προς την προτινόμενη λύση. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει, πρέπει να συνεχιστεί η διαβούλευση, να συζητήσουμε τις διάφορες προτινόμενες λύσεις και να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Άλλοι συνάδελφοι είπαν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Και βέβαια, τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν μεταξύ τους, αντιμετωπίζουν διαφορετικές καταστάσεις. Ωστόσο, εμείς εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ λύσεις. Και θα πρέπει να προτείνουμε τόσο νομοθετικά όσο και μη νομοθετικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν τα εντοπισμένα αυτά προβλήματα. Να τονίσω επίσης αυτά που μας είπε η κυρία Στόλα όσον αφορά την δημόσια διαβούλευση. Μας είπατε ότι είναι 77% των συμμετεχόντων στη διαβούλευση μας είπαν τελικά ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε νέες λύσεις για την εξορρόπηση επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Μα αυτό από μόνο του σημαίνει ότι εμείς ως όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επιγόντως να βρούμε τη λύση αυτή, μόλον ότι το όλο εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Πρέπει λοιπόν εδώ εμεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να καταλήξουμε σε μια λύση, να προτείνουμε αν μη τι άλλο μια λύση. Πρέπει η κατάσταση να αλλάξει επιγόντω. Ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει επίσημε προτάσει μέχρι τα τέλη του έτου ή έστω μέχρι τι αρχέ του επόμενου έτου, προκειμένου να έχουμε επιτέλου στα χέρια μα ένα έγγραφο συγκεκριμένο το οποίο θα μπορέσουμε να αναλύσουμε, να τροποποιήσουμε και εν τέλει να εγκρίνουμε προκειμένου να βρούμε μία λύση. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω σε ένα επικοδομητικό διάλογο και στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Πλίνκεβιτσιούτε, η συγγήτρια της Επιτροπής ΦΑΜ και δίνω τώρα ε, τον λόγο στην κυρία Στανόκα που είναι η συγγήτρια για την Επιτροπή Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους επικεφαλείς των Γενικών Διευθύνσεων και τους συναδέρφους. Οι περισσότερες παρατηρήσεις σας ήταν θετικές. Προσβλέπουμε στις περαιτέρω προτάσεις σας. Μας περιόριζε κάπως ε, το μήκος της έκθεσης. Συνεργαζόμαστε τώρα με τους σκιώδες, σκιώδες ώστε να συμπεριλάβουμε όσο γίνεται περισσότερες προτάσεις. Οι επικρίσεις που ακούστηκαν συνδέονταν κυρίως με την αρχή της επικουρικότητας. Μιλάμε όμως όχι μόνο για νομοθετικές προτάσεις, αλλά και για μη νομοθετικές προτάσεις. Θα πρέπει να συνδυάσουμε λοιπόν και τις μεν και τις δε, έχοντας πάντα κατά νου την επικορικότητα. Θέλουμε να πετύχουμε σύγκληση της κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη. Και οι δύο εισηγήτριες προερχόμαστε από νέα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα ε, χώρες της Βαλτικής και η δική μου χώρα, η Λετωνία, έχει εφαρμόσει την οδηγία για την γονική άδεια χωρίς προβλήματα. Αλλά μας ενδιαφέρει το θέμα και της άδειας πατρότητας. και θα χαρούμε πολύ να δούμε σχετική νομοθετική πρόταση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε όλους και ελπίζω να συνεχίσουμε την επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα θυμάστε ότι η πρώτη κοινή μα ε, συνεδρίαση για το θέμα αυτό ανάμεσα στι Επιτροπές ε, Απασχόλησης και Γυναικών ε, πραγματοποιήθηκε την ημέρα των βομβιστικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες και αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη συνεδρίαση. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα είχαμε χρόνο να κάνουμε τη συζήτηση και είμαι βέβαιη ότι θα βρούμε λύσεις ώστε να πετύχουμε και πλειοψηφία ε, στην Ολομέλεια. Προθεσμία την υποβολή τροπολογιών είναι η 30 Μαΐου. Εξέταση των τροπολογιών θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Απασχόλησης 16 Ιουνίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών στις 12 Ιουλίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο, μετά το καλοκαίρι δηλαδή. Νομίζω ότι πετύχαμε το στόχο που θέλαμε. Να περιμένουμε να δούμε τώρα λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Και σας ευχαριστώ ε, που είχαμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση.